Herr Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Παρακαλώ, αγαπητέ κυρίε και κύριοι, να καθίσετε. Κυρίε και κύριοι, σε δύο αλλεπάλληλε βομβιστικές επιθέσεις, εκρήξεις μάλλον εχθές ε, στη Βοστόνη έχασαν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι και πολύ περισσότεροι τραυματίστηκαν σοβαρά. Ε, μια αθλητική εκδήλωση ο Μαραθώνιος της Βοστόνης στον οποίο ε, συμμετέχουν άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο σε μια πόλη η οποία συμβολίζει όσο καμία άλλη τον αγώνα για την ελευθερία. Εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνω τα θερμά μας ε, συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και εύχομαι ταχύτατη ανάρρωση στους τραυματίες. Θα ήθελα να απευθύνω επίση θερμένη ευγνωμοσύνη προ τι αρχέ των ΗΠΑ και τι ομάδε διάσωση και καθώ παραμένει ακόμη αδιευκρίνηστο ποιο τοποθέτησε και πυροδότησε του κριτικού μηχανισμού, πρέπει να πω με κάθε σαφήνεια ότι η τρομοκρατία ποτέ δεν έχει δικαιολόγηση και βρισκόμαστε στο πλευρό των Αμερικανών φίλων μα. Οι σκέψει ε, οι σκέψεις μας είναι κοντά τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.